Οι αρμόδιε πολεωνικέ αρχέ μου έχουν διαβιβάσει μια αίτηση άρση τη ασυλία του κυρίου Γιάννη Κόρβιν Μίκε βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να παραπευθεί στη νομική επιτροπή του Κοινοβουλίου που είναι και